Καλημέρα σε, σε όλους και εσείς που είστε εδώ και όλοι βρίσκεστε κάπου στην ε, Ευρώπη. Έχουμε αυτή την ε, έκτακτη κοινή συνεδρίαση Επιτροπής Προπολογισμών και Οικονομικής Επιτροπής ε, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και φαντάζομαι ότι εγκρίνεται την ημερησία διάταξη και ότι δεν υπάρχουν ε, προτάσεις ε, αλλαγών, οπότε να σας ε, ξεκινήσω την εισαγωγή μου για την γίνημα συνεδρίαση και καλώς όρισαν τέσσερις ομιλητές μας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Άντριο Μακντάουελ, ο εκτελεστικός διευθυντής Βίλεν Μόλτερερ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Σωτικών Επενδύσεων, ο διευθύνων σύμβουλος, ο σύμβουλος του Ταμείου Παρακρατικών και Δαμείων Φαμπρίτσιο Παλέρμο και επίσης ε, ο διευθυντής του οργάνωσης Αντίβαρο, Ξαβιέ Σόλ. Και επίσης ε, όλοι οι συνάδελφοι καλωσόρισαν. Ο σκοπός της ακροασής μας είναι να συζητήσουμε ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει ο, ο όμιλος ε, της ΕΤΕ σε σχέση με το να αποκτήσουμε ανθεκτικότητα στα υγειονομικά και στα επιχειρηματικά κατόπιν της πανδημίας και της φάσης Τη ανάκαμψη. Οπότε κατευθείαν να πάμε στο κεντρικό μας θέμα. Τα τελευταία δεδομένα πληροφορίες για τον Μάρτιο από την Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι οι αποταμιεύσει των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά σε όλη την Ένωση μετά την ε, πανδημία. Και επίση έχουμε κάποια πρώτα δεδομένα για την περίοδο μέχρι τα μέσα Μαΐου που φαίνεται ότι αυτή η αύξηση του ρυθμού των ε, των, των, των, των αποταμιεύσεων ε, όσο προχωρούσε η κρίση ε, γινόταν πιο έντονη, αυξανόταν. Και αν, έχουμε ε, αν δεν έχουμε μάλλον κάποιο πίσω γύρισμα, κάποια αντιστροφή αυτών των τάσεων και αν έχουμε χαλάρωση σημαίνει ότι, ότι τα περιθώρια όσον αφορά την ανάκαμψη ίσως είναι μικρότερα ε, σε σχέση με το παρελθόν. Άλλη ε, δυνατότητα, πιθανότητα είναι να μπορέσουμε να έχουμε κάποια ανάκαμψη βάση εξαγωγών αλλά βλέπουμε ότι έχουμε συρρήγνωση της ε, παγκόσμιας οικονομίας, 3% σύμφωνα με το δου, του και βλέπουμε ότι αυτή η ατμομηχανή των εξαγωγών δεν θα βοηθήσει και πάρα πολύ όσον αφορά την ανάκαμψη. Επομένως, ε, θέλουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να μετέλθουμε ούτω ώστε να βοηθήσουμε την οικονομία της Ένωσης και βέβαια μετά την κατανάλωση και εξαγωγές έχουμε τις επενδύσεις. Εδώ λοιπόν μπαίνει το θέμα του ρόλου της ΕΤΕ. Το θέμα ε, δεν είναι το πότε αλλά το με ποιο τρόπο. Τι μέσα μπορούμε ε, να μετέλθουμε και να ανακατευθύνουμε ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στο προβλήματα ε, τα οικονομικά από την πανδημία και πώς είναι δυνατόν αυτά τα νέα μέσα πολιτικής να μας δώσουν την επιθυμητή όθηση για την οικονομία της Ένωσης και για αυτό ε, το Eurogroup της 15ης Πέμπτου συζήτησε τα σχετικά με την πανευρωπαϊκή εγγύηση, αυτό το δίκτυο ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, το οποίο θα το υλοποιήσει η ΕΤΕ και θα πρέπει να ενημερωθούμε περισσότερο για τις παραμέτρους αυτής της κίνησης και τη διαχείριση κινδύνου, οπότε βέβαια πάντοτε η πολιτική σημαίνει επιλογές, σημαίνει ότι κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις και ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα βοηθήσει να δούμε τι θα κάνει η ΕΤΕ όσον αφορά τη διαδρομή που έχουμε μπροστά μας. Και τώρα να δώσουμε τη σκητάλη στην ε, συμπρόεδρο, την Ιρένε, η κυρία Τινάλια, η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έρχομαι και εγώ τώρα στη συνεδρίαση. Καλώς όρισαν οι ομιλητές μας για αυτή την ε, από απόσταση ακρόαση. Ο ρόλος της ΕΤΕ είναι πάρα πολύ σημαντικός όσον αφορά τις ε, επενδύσεις παντού, παντού αυτό τα περισμένα χρόνια και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μας εξηγήσουν οι ομιλητές μας την ε, εμπειρία τους όσον αφορά τα μέχρι σήμερα χρησιμοποιημένα μέτρα πολιτικής όπως το πρόγραμμα ΕΦΣΙ όπως ε, ανέφερε συμπρόεδρε και για το τι άλλα μέσα έχουμε για να ανασχέσουμε τις συνέπειες της πανδημίας και να προχωρήσουμε στην ανάκαμψη. Να δούμε, έχουμε αυτή η χαλάρωση για τις κρατικές ε, επιχορηγήσεις, έτσι θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις από τα κράτη και βέβαια έτσι θα βοηθούν και οι εργαζόμενοι, αυτό είναι μια ευκαιρία και θα πρέπει να δούμε το ότι ε, υπάρχουν αποκλήσεις ε, θα βοηθήσουμε την κοινή, την ενωμένη στην ενιαία αγορά, συγγνώμη, ακούγεται πολύ άσχημα η ομιλήτρια. Οπότε, να δούμε το πώς θα αναδειχθεί πιο ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την υπόθεση. Και πάλι σας ευχαριστούμε των προτέρων τους ομιλητάς. Irene, σε ευχαριστούμε. Λέει ο κύριος Όφερτβελτ. Τώρα για να δούμε πώ θα γίνει η διαδικασία για την ακρόασή μα. Ο καθένα από του τέσσερι προσκεκλημένου πρόκειται να έχει 7 λεπτά τόσο ώστε να κάνει την εισαγωγή του και αυτό πρόκειται ε, στη συνέχεια ε, να συνεχιστεί με ερωταπαντήσεις από τις δύο επιτροπές μας ε, δύο λεπτά κάθε ερώτηση και κατόπιν θα έχουν οι προσκεκλημένοι 8 λεπτά για να απαντήσουν οπότε σας παρακαλώ να σεβαστείτε αυτό το χρονικό όριο όσο μπορείτε περισσότερο γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης και έχουμε διερμηνία από γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά. Οπότε, αρχίζουμε τώρα του τους ε, προσκεκλημένους μας. Όμω, θα πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά με τον οποίο θα μιλήσουν, γιατί έχουν κάποια προβλήματα ε, σύνδεση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μακντάουλ, μετά ο κύριο Μόλτερ, μετά ο κύριο Παλέρμο. Ε, θα αρχίσουμε επομένω ε, με τον κύριο Παλέρμο. Έχετε το λόγο, κύριο Παλέρμο. Λέει, αυτή θα είναι η καινούργια σειρά. Με μεγάλη μου χαρά ε, βρίσκομαι εδώ, κυρίε και κύριοι. για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να ως ΕΤΕ να κάνουμε κάτι για την πανδημία. Πρώτα πρώτα που ξέρουμε έχουμε το Ίδρυμα CDP, το οποίο υπάρχει εδώ και 170 χρόνια και η αποστολή του είναι η εξή στην Ιταλία. Να υποστηρίξει την οικονομία, να μπορέσει να αξιοποιήσει τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια ε, των 27 εκατομμύριων Ιταλών, να βοηθήσει για απασχόληση και ανάπτυξη. Σήμερα ε, αποτελούμε έναν όμιλο που έχει ενεργητικό περίπου 450 δις όσον αφορά αυτές τις ε, καταθέσεις και 34 δις επίσης ε, σε μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης θέλαμε να ενεργοποιήσουμε από το 2018 ένα business plan για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη στη χώρα και τώρα έχουμε επικεντρωθεί στα εξή τρία μέτωπα, καινοτομία, βιωσιμότητα και ε, δράση ε, επιτόπου. Δηλαδή στην επικράτεια της Ιταλίας για την καινοτομία έχουμε αυτό το ταμείο, το οικοσύστημα για να μειώσουμε την απόσταση και ε, επομένως έχουμε αυτό το ταμείο της καινοτομίας επαναλαμβάνω και όσον αφορά την βιωσιμότητα, ξεκινήσαμε επίσης ε, κάποια σχέδια, προγράμματα τα τελευταία χρόνια για την κυκλική οικονομία και ανανεώσιμη ενέργεια. Όσον αφορά κάποιες στρατηγικού χαρακτήρα εταιρείε και όλα αυτά εκτίθενται στη σχετική μας έκθεση. Αυτό το οποίο θέλουμε τώρα ε, από πρακτική άποψη είναι να έχουμε πιο έντονη παρουσία και να έχουμε καλύτερη επαφή με τους ε, ομολόγους μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα καινούργια γραφεία. Ε, Επίση καινούργια υπηρεσία δική μας για τις υποδομές. Να βοηθήσουμε δηλαδή την κυβέρνηση ούτω ώστε να σχεδιάσει τις επενδύσεις στις υποδομές. Οπότε το Ταμείο Παρκατικών και Δανείων είναι σε επαφή με τους ομολόγους μας σε όλη την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχουμε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να συνεχιστεί αυτή η δέουσα συνεργασία. Η συνεργασία έχει υπάρξει πάρα πολύ αποδοτική να θέλουμε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ, να χρηματοδοτήσουμε τα έργα υποδομής, αλλά και την καινοτομία. Στα πλαίσια αυτής της πανδημίας χωρίς προηγούμενο, το Ταμείο μας έχει εξαγγείλει κάποιες πρωτοβουλίες. Όπως τα γνωρίζετε. Έχουμε προχωρήσει σε μέτρα για περισσότερη ρευστότητα, για καλύτερη πρόσβαση στην δανειοδότηση, για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρείε. Τρία δις διατέθηκαν και σύντομα θα έχουμε από την ΕΤΕ άλλο 1,5 δις. Επίσης, διευκόλυνση δανειοδότησης προς εταιρείε και για ε, επίσης για τις ε, εταιρείε τύπου mid-caps αλλά και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, τώρα διαπραγματευόμαστε 34 δις δανείων και επίσης πρόκειται έτσι να βοηθήσουμε κατά 1,4 δις δήμους και κοινότητες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνέργειες με την ΕΤΕ και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα ε, θα πρέπει να διαπιστώσω ότι οι σχέσεις μας με τον Όμιλο ΕΤΕ είναι ισχυρή και προσωδοφόρα. Έχουμε επίσης για καινοτομία, για υποδομές και για ΜΜΕ ε, το πλάνο Juncker. 9,4 δις ε, είναι η πρικοδότηση των τεσσάρων πλατφορμών επένδυσης που έχουμε. Επίσης, για έρευνα και ανάπτυξη έχουμε ε, κάποια προγράμματα και έχουμε αποσπάσει αποτελέσματα. Θέλουμε για τις ΜΜΕ να ενεργοποιήσουμε τέσσερις πλατφόρμες με 14 δις για ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας και επίσης σε συνεργασία με την ΕΤΕ ε, θέλουμε να βοηθήσουμε και για τις θεομηνίες ε, και έχουμε διαθέσει τρία δις για την ρευστότητα. Όμως θέλουμε να υπάρχει εξυγχρονισμός των σχολείων στην Ιταλία. Μόχλευση από πλευράς της ΕΤΕ. Οπότε με την ΕΤΕ ήταν πολύ αποδοτική συνεργασία και για mid-caps έχουν δοθεί κάποια δισεκατομμύρια και επίσης μια γραμμή εγγύησης για τις μικρές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο και πρώτα-πρώτα να υπάρχει ανταγωνιστική χρηματοδότηση για τις NPI και θέλουμε επίσης με αυτούς τους ε, πόρους να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία και αυτές οι εθνικές ε, επιχειρήσεις να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Τώρα, η χρηματοδότηση αυτών των εθνικών ε, NPIs συνήθως είναι υψηλό. Και το θέμα αφορά τις χώρες που δεν έχουν τριών 3α. Οπότε θέλουμε να υπάρχει όλο ένα και περισσότερη στήριξη από την ΕΤΕ στους εθνικούς εταίρους. Γι' αυτό το 1,5 δις από πλευράς της ΕΤΕ για την ρευστότητα είναι ένα μέτρο πολύ θετικό. Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι μόνο ένα πρώτο βήμα όσον αφορά και περαιτέρω μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Δεύτερον, σε σχέση με τις τοπικούς φορείς και εταιρείε θεωρούμε ότι μπορούμε να τους δώσουμε τους πόρους που χρειάζονται και υπάρχουν. Και σε αυτό θα βοηθήσει η πρόσβαση σε κάποιες εγγύησεις από το Invest EU. Οπότε θέλουμε καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις στους δυναμικούς τομείς και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε ε, κάλυψη και των ε, μη προνομιούχων περιοχών της χώρας μας όπως η κεντρική και η νότια Ιταλία και εκεί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά ε, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε τις τοπικές διομορφίες και σας ευχαριστώ. Α, γιατί πιστεύουμε πάντως ότι μπορεί αυτή η κρίση να γίνει μια ευκαιρία και η ΕΤΕ να βοηθήσει περισσότερο με καλύτερη συνεργασία. Να βοηθήσει στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το Ταμείο μας και εγώ προσωπικά θα παλέψουμε για την επιτυχία αυτής της διαδρομής. Σας ευχαριστώ και περιμένω τις απόψεις. On Περιμένουμε ακόμη να αποκατασταθεί η σύνδεση με τους κυρίους Μακδάουελ και Μόλτερερ. Γι' αυτό θα έλεγα να περάσουμε τώρα στον κύριο Χαβιέρ Σόλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Σόλ, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση. Με τιμά ιδιαίτερη παρουσία μου σε αυτό το πάνελ με τόσο α, α, κορυφαίους καλεσμένους. Είμαστε ένα συνασπισμός από εννέα με κυβερνητικές οργανώσεις που θέλουμε να καταστήσουμε την, α, τα ευρωπαϊκά δημόσια οικονομικά κινητήριο δύναμη προς τη μετάβαση σε κοινωνίες κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες και δίκαιες. Ε, από αυτή την άποψη παρακολουθούμε δραστηριότητες της ΕΤΕ ευαίσθητα θέματα όπως είναι δραστηριότητες ε, μέσω φορολογικών παραγόντων, ε, φορολογικών παραδείσων ή στηρίζοντας ορυκτά καύσιμα και είμαστε υπέρ βαθύτατων μεταρρυθμίσεων στην ΕΤΕΠ. Οπότε θέλουμε να συμμετέχει η ΕΤΕΠ και να αναδειχθεί ο ρόλο της ε, στο πακέτο ανάκαμψης, αλλά με κάποιες, ε, με λήψη υπόψη των βασικών προκλήσεων και των συστάσεών μας. Καταρχήν, ε, η βασική μας παρατήρηση είναι ότι η ΕΤΕΠ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα συνεχίσει το μετασχηματισμό της σε μια τράπεζα για το κλίμα, περνώντας σε μια πιο δημοκρατική διαφανή ε, και βιώσιμη δομή ή θα κρατήσει την πολιτική μία από τα ίδια και θα χάσει μια ιστορική ευκαιρία να θέσει και ένα προηγούμενο μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών έχει ένα εμβληματικό ρόλο λοιπόν στη δεσμή μέτρων ε, για την ανάκαμψη. Ήδη οι εμπορικέ τράπεζε έχουν λάβει πολύ ε, ρευστότητα για να αντιμετωπίσουν την κρίση και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΤΕΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ιδιαίτερο έργο τη. Να προωθήσει τι ε, επενδύσεις και να στηρίξει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, κυρίως και μεταξύ άλλων και αυτές που έχει θέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λαμβάνοντα υπόψη όμω και αποδεικνύοντα την προσεδικότητα αυτών των επενδύσεων. Η ΕΤΕΠ δεν είναι μόνο τράπεζα, είναι μια δημόσια τράπεζα, είναι ο χρηματοοικονομικός τη Ευρωπαϊκή Ένωση. με μια δημόσια και μακροπρόθεσμη αποστολή. Και οι επενδύσει τη ΕΤΕΠ είναι κυρίω μακροπρόθεσμα δάνεια, όχι επιδοτήσει. Οπότε ο ρόλο που θα διαδραματίσει η ΕΤΕΠ στην οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να θεωρηθεί υπό αυτό το μακροπρόθεσμο πρίσμα και προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε κέρια σημασίας να εξασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕΠ δεν θα επιδεινώσουν τις κοινωνικές ανισότητες και την έκτακτη κατάσταση για το κλίμα και το περιβάλλον και θα προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους και τις μικρές επιχειρήσεις και όχι αυτούς που ήταν υπέτη για το ότι οι κοινωνίες μας έχουν καταντήσει να είναι τόσο εύθραυστες. Πρώτον, το στόχος της υιοθέτηση ε, του οδικού χάρτη για το κλίμα, τον οποίο επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μέχρι το 2020, ο στόχος αυτός θα πρέπει να παραμείνει. Η ΕΤΕΠ θα πρέπει να θετήσει μια φιλόδοξη στρατηγική ώστε να μετατραπεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα του Κλίματος και να ε, χαράξει το μακροπρόθεσμο ρόλο της ΕΤΕΠ κατά την καθοδήγηση των οικονομιών προς ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μονοπάτι. Επίσης, οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι αντικυκλικές και να μην τροφοδοτούν σχέδια και επιχειρήσεις που αντιβαίνουν στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Ε, οι επενδύσεις ε, με μακροπρόθεσμα και μη βιώσιμα αποτελέσματα θα πρέπει να αποφεύγονται. Ε, ισχυρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και η αρχή του μη βλάπτην θα πρέπει να αποτελούν τη βάση όλων των ε, δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ και στα πλαίσια της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη, αλλά και για το σύνολο του χαρτοφυλακίου του ομίλου ΕΤΕΠ. Δεύτερον, θεωρούμε κρίσιμο να θέσει όρους στη χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ, ώστε οι εταιρείε που θα στηρίζονται από τα νέα μέτρα και από το νέο Ταμείο Εγγύσεων θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και μελλοντικέ κρίσει. Και η ΕΤΕΠ θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να απαγορεύσει ε, εταιρείε που λαμβάνουν την, ε, την στήριξη της ΕΤΕΠ να καταβάλουν μερίσματα στους ε, μετόχους, να δίνουν πρίμα στους γενικούς διευθυντές ή να πραγματοποιούν επαναγορά ιδίων μετοχών. Θα πρέπει να αναγκάσει τις εταιρείες να προστατεύσουν τους εργαζομένους τους και να εξασφαλίσουν θέσεις απασχόλησης προσφέροντας αξιότυπες, αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες. Επίσης, θα πρέπει να, να απαιτεί από τι ε, μεσέ και μεγάλε επιχειρήσει ένα αξιόπιστο σχέδιο για αποαθρακοποίηση των δραστηριοτήτων τη, προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Γενικώ, ε, τα λάθη του παρελθόντο ε, δεν θα πρέπει να επαναληφθούν. Λάθη που συνέβαλαν στο να γίνουν πιο τρωτέ οι κοινωνίε κατά την αντιμετώπιση τη κρίση, όπω η χρηματοδότηση τη ιδιωτικοποίηση ουσιοδών δημοσίων υπηρεσιών. Αυτά τα λάθη λοιπόν θα πρέπει να αποφευθούν. Και εδώ είναι μεγάλη ευθύνη τη ΕΤΕΠ γιατί στο παρελθόν δρομολόγησε τεράστια δημόσια κονδύλια για να στηρίξει ε, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα στην Ιταλία και την Ιρλανδία. Είναι λοιπόν ε, ένα σημείο καμπής για τα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως χρηματοοικονομικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θέσει μια μακροπρόθεσμη πορεία. Από τη μια συμβάλλοντας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και σε μια δίκαιη μετάβαση αντιμετωπίζονται τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν περιφέρειες και κοινότητε που ήδη υστερούν, που ήδη έχουν μείνει πίσω και πασχίζουν να πραγματοποιήσουν αυτή την πράσινη μετάβαση. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει η ΕΤΕΠ να γίνει πιο διαφανέ ε, και δημοκρατικό όργανο, δημόσιο ε, οργανισμό, προκειμένου να υλοποιήσει τη δημόσια αποστολή εξυπηρετώντα του Ευρωπαίου πολίτε και τι ευρωπαϊκέ περιφέρειε. Και από αυτή την άποψη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην αποκατάσταση τη ε, Διαφάνεια και τη λογοδοσία τη ΕΤΕΠ, στην ενίσχυσή τη. Πρόσφατα είχαμε κάποιε αποκαλύψει στου Times του Λουξεμβούργου που επιβεβαιώνουν κάποια επικριτικά μα συμπεράσματα. Προ το παρόν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τον έλεγχο των κονδυλίων τη ΕΤΕΠ. Ε, Ελλειπή, για παράδειγμα, δέουσα επιμέλεια στην επιλογή των πελατών ή στην προβληματική αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης και διαφθοράς. Εν κατακλείδη, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε τα σχέδια ανάκαμψη ΕΤΕΠ να αποφεύγουν τη Γιάννη, τη πάντα, μία από τα ίδια, και να εξασφαλίσουν περισσότερες επενδύσεις σε μια οικονομία ουδέτερη από άποψη άνθρακα, προσφέροντα κοινωνική προστασία σε κοινότητες που έχουν πληγεί από αυτή την απανθρακοποίηση. Επίσης, θα πρέπει τα σχέδια ανάκαμψη να είναι διαφανή για του πολίτε. Και αυτό είναι σημαντικό καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί σε τελική ανάπτυξη, σε τελική ανάλυση, αν έχουμε πραγματικά δημοσιονομικά δίκαια οικονομικά, θα έχουμε μια, ένα πραγματικό δυνητικό δυναμικό για την καθοδήγηση τη οικολογική μετάβαση, αντιμετωπίζοντα τι κοινωνικέ ανισότητες και βελτιώνοντα τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των κοινωνιών μα. Σα ευχαριστώ και είμαι έτοιμο να απαντήσω σε ερωτήσει σα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλ. Από ό,τι φαίνεται λύσαμε το πρόβλημα της σύνδεσης με τον κύριο Μόρτερερ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, ωραία, οπότε με τα χαράς να του δώσω το λόγο. Κύριε Μίλαν Μόρτερερ, έχετε το λόγο. Αν ο κύριος Μόρτερερ πατήσει το κουμπί που λέει speech, speak, με ακούτε? Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που προσπάθησαν οι υπηρεσίες ε, να το λύσουν ε, και για τον Αντιπρόεδρο Μακντάουλ. Κρίμα που εγώ έλυσα το πρόβλημα πρώτα και θα μιλήσω πριν από τον Αντιπρόεδρο που θα ομιλήσει εκ μέρους του ομίλου. Οπότε εγώ θα περιοριστώ στο να μιλήσω ως εκτελεστικός διευθυντής του ΕΦΣΥ. Κυρίες και κύριοι, μετά την τελευταία μας ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018, πολλά έχουν μεσολαβήσει και θέλω να σας ευχαριστήσω που σήμερα μου δίνετε τη δυνατότητα να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την ανταπόκρισή μας στην κρίση της COVID-19. Θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντας σε όλους μας το γεγονός ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο ψήφισε στα τέλη του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Πρόκειται καταρχάς για τη βελτίωση του ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου. Κατά δεύτερον υπάρχει ο συμβουλευτικός πυλώνας που έχει μεγάλη σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και το τρίτο σκέλος είναι το χρηματοοικονομικό για τις στρατικές επενδύσεις. Το 2018 ήταν ένα κρίσιμο έτος για αυτό το Ευρωπαϊκό Τέμιο Στρατηγικών Επενδύσεων. Όπως γνωρίζετε, ελήφθησαν το 2018 τέσσερις σημαντικές αποφάσεις. Η πρώτη αφορούσε την παράταση ε, της ισχύω ε, του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2020 και την αύξηση του όγκου και των στόχων. Έπειτα, με 500 δις. Έπειτα, προσθετικότητα, δηλαδή προσθέμενη αξία. Τρίτον, ένας νέος στόχος τέθη, ο κλιματικός συγκεκριμένο στόχος, με πρόθεση οι επενδύσεις που σχετίζονται με το κλίμα να ανέρχονται στο 40% στο πλαίσιο του παραθύρου ε, υποδομών και καινοτομίας. Και επίσης υπάρχει το λεγόμενο σκεπτικό ή πίνακας επιδόσεων. Θα σας κάνω μία επισκόπηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά διακόπικη σύνδεση. I'm looking at the technical Ο πρόεδρος, στρέφομαι στους τεχνικούς μας. Mr. can you... Ο κύριος Μόλτερερ μπορεί να πατήσει ξανά το κουμπί Speak. Βλέπουμε αλλά δεν ακούμε τον κύριο Μόλτερερ. Mr. Δεν ακούμε τον κύριο Μολτερέρο. Ε, Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο προφανώς στο μιλητή. Όπως λέει και ο τεχνικός. Mm, mm, we cannot hear you. Can you, Κύριε Μόλτερ, δεν σας ακούμε. Μπορείτε να κάνετε ένα refresh, μια ανανέωση της σελίδας σας, παρακαλούμε. Μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του iPad, κύριε Μόλτερερ. Παρακαλούμε, κάντε το αν έχετε την καλοσύνη. Mr. McDowell, we see you are connected. Βλέπω ότι ο κύριος Μακντάουλ συνδεθεί αν θέλει να πάρει το λόγο στο μεταξύ. Παρακαλώ πατήστε το κουμπί speak κύριε Μακντάουελ. Nothing? Uh, Τίποτα. Από ό,τι φαίνεται και οι δύο μιλητές έχουν πρόβλημα. Είναι συνδεδεμένοι, μπορούν να μας ακούσουν, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Οπότε, προτείνω να ακούσουμε τους ε, βουλευτές τα μέλη της Επιτροπής ε, Προεπολισμών και τα μέλη της Επιτροπής της Οικονομικής. Ελπίζω στο μεταξύ να βελτιωθούν οι συνδέσεις των δύο ομιλητών για να μπορέσουν έστω τις ερωτήσεις σας να απαντήσουν αφού τις ακούσουν. Μας ακούνε, να μου το επιβεβαιώσετε παρακαλώ ότι μας ακούν. Διότι αλλιώς ε, είναι και λίγο παράλογο να κάνουμε ερωτήσεις σε κάποιον που δεν ακούει. Κύριε Μόλτερ, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί speak. Βλέπω ότι συνδεθήκατε ξανά. Ο κύριος Μόλτερ ακούγεται. Μπορώ να συνεχίσω, λέει ο κύριος Μόλτερ. Βεβαίως, κύριε Μόλτερ, μπορείτε. Να σας επισημάνω ε, κάποια πράγματα σε σχέση με το που βρισκόμαστε. Ε, ο Όμιλος είναι ε, η ΕΤΕΠ και το Ταμείο έχουμε περίπου 89,9 δις χρηματοδότηση με βάση την εγγύηση. Ε, ελήφθησαν οι αποφάσεις ε, που πλέον έχουμε 486 δισεκατομμύρια κινητοποιημένες επενδύσεις σε σχέση με το στόχο των 500 δις όλα τα κράτη-μέλη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, Εσείς ε, μιλήσατε για αυτό το στόχο 40% για την κλιματική δράση. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στο 42% στο ότι αφορά το σύνολο των ε, επενδύσεων σε αυτό το παράθυρο υποδομών και καινοτομία, που σημαίνει ότι είμαστε μέσα στο στόχο μας και έχουμε αυξήσει και το μερίδιο των ε, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κλίματος κατά 6% μέχρι τώρα. Άρα και πάλι είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σε, καλή, ε, σε καλό δρόμο. Σε ό,τι αφορά τους τομείς, βασικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτοί έχουν ωφεληθεί περισσότερο. 30% του συνόλου των επενδύσεων ε, του ομίλου που στηρίζονται από, το, ε, από την εγγύηση του ΕΦΣΗ, χρηματοδότησαν ΜΜΕ. Δεύτερη κατηγορία περίπου 26% και με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό που μπορώ να σας το αναφέρω, είναι η έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, άρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη. Και τρίτη προτεραιότητα, ενέργεια, δηλαδή ανανόσιμε πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, υποδομές. Οι υποδομές εδώ ανέρχονται περίπου στο 17%. Άρα και εδώ είμαστε σε, καλή, ε, σε καλό δρόμο ό,τι αφορά τους στόχους και σε σχέση με τους τομείς που είχαμε από την αρχή ε, εστιάσει. Να σας δώσω κάποια στοιχεία ε, για τη γεωγραφική κατανομή. Πάνω από 4 στα 10 έργα εύση απευθύνονται άμεσα σε περιοχές συνοχής. Ονομαστικά τα στοιχεία θα σας δείξουν ότι οι τρεις μεγαλύτερες χώρες ευσύ είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτό δεν σας εκπλήσει λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των οικονομικών χωρών αυτών. Αν όμως συσχετίσουμε τις επενδύσεις με το ΑΕΠ, τότε η εικόνα αλλάζει εντελώ. Και βλέπουμε ότι οι πέντε βασικοί δικαιούχοι, ε, χώρες που έχουν ωφεληθεί δηλαδή, είναι η Ελλάδα, η Εστονία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Ισπανία. Ακριβώς δηλαδή αυτές οι χώρες και περιοχές που είναι και στο επίκεντρο ε, της δράσης μας. Κάτι πολύ ενδιαφέρον και βασικό χαρακτηριστικό του ΕΦΣΙ είναι ότι το 25% περίπου όλων των επενδύσεων βασίζονται στη συνεργασία με εθνικές ε, τράπεζες ή άλλους οργανισμούς προώθησης, promotional banks. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η συνεργασία δηλαδή με τέτοιους οργανισμούς που πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής και βλέπω ένα τεράστιο δυναμικό. Για να σας δώσω συγκεκριμένα νούμερα, πάνω από 1,1 εκατομμύριο ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επωφεληθεί από την εγγύηση αυτού του Ταμείου Εγγύησεων μόνο και μόνο από το Ταμείο Εγγύησεων. Και ιδίω αν λέω και τους ε, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά την ανανεώσιμη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 10 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου έχουν ωφεληθεί από επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια. 33 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου ωφελούνται από έργα στον τομέα της επεξεργασίας λιμάτων και της κυκλικής οικονομίας και Έχουμε 500.000 περίπου ε, προσιτά ε, από οικονομικής πλευράς διαμερίσματα, τα οποία είτε ε, τίστηκαν είτε ανακαινίστηκαν. Επίσης, το οικονομικό τμήμα, σε μακροοικονομικό επίπεδο τώρα, έκανε μία μελέτη με βάση το μοντέλο Ρόμελο και μας λένε ότι υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που υποστηρίχθηκαν με την εγγύηση εύση και 1,9% προστέθηκε στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ή θα προσθεθεί μέχρι το 2022. Άρα και από μακροοικονομικής πλευράς ε, είναι πολύ καλές επιδόσεις μας. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω πως μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους θα έχουμε πετύχει το στόχο των 500 δις. Μπορώ να σας το πω και να σας το υποσχεθώ κιόλα. Αφού είμαστε ήδη στα 486. Επίσης τα πάμε πολύ καλά και με τους πολλαπλασιαστές. Το crowding in. Πάει καλά και εδώ το πράγμα. Όπως προβλέπω ο κανονισμός, από το 2008 έχουμε το scoreboard και το rational ε, τον πίνακα επιδόσεων και το σκεπτικό για τις αποφάσεις μας. Εκτός βέβαια αν υπάρχουν κάποια θέματα εμπορικού απορρίτου. Οπότε τα στοιχεία γίνονται, δίνονται στη δημοσιότητα μετά την υπογραφή. Να πω ότι το ΕΦΣΙ στηρίζει γενικά ε, τις επιχειρήσεις αλλά και ε, εν μέσω κρίσης COVID. Θα σας πω ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες μας. Στηρίζουμε γιατί υπάρχει αυξηνόμενη ζήτηση. Στηρίζουμε λοιπόν τη δανειοδότηση των ΜΜΕ μέσω ε, των εγγύσεων Έχουμε μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση στην Επενδυτική Επιτροπή σε σχέση με αυτέ τι δραστηριότητε. Η Επενδυτική Επιτροπή ήταν έτοιμη μάλιστα να επιταχύνει και την όλη διαδικασία για να μπορούμε να αντιδράσουμε πιο γρήγορα. Δεύτερο σκέλο, δεύτερο άξονα, αύξηση τη χρηματοδότηση και της υποστήριξης ε, στα υφιστάμενα έργα και σχέδια. Πρέπει να τους χάρη ε, επενδύσει υποδομών στον τομέα της υγείας. Τρίτο σκέλος, τρίτος άξονας. Στήριξη στον τομέα της έρευνας καινοτομίας και ανάπτυξης, ε, RDI. Από την αρχή είπα ότι αυτός είναι ένας από τους πυρήνες επιτυχίας ε, της ε, δράσης μας στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. 37 ε, υψηλά ε, εξειδικευμένε σε τεχνολογίες εχμής εταιρείε μεσαία κεφαλαιοποίηση έχουμε υποστηρίξει μέχρι τώρα και περιμένουμε πολύ περισσότερα τέτοια επενδυτικά ε, προγράμματα να προχωρήσουν. Ολοκληρώνοντας, ε, μπορώ να σας πω ότι το ΕΦΣΙ είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει αξιοποιώντα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρηματοδοτικά μέσα που έχει στη διάθεση το όμιλος ε, της ΕΤΕΠ που είναι το οικονομικό σκέλος και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που παρέχει την εγγύηση. Δεύτερον είναι και πολύ αποτελεσματική στη συγκέντρωση ιδιωτικού κεφαλαίου, ο παλαπλασιαστή λειτουργεί, όπως είπα, και τρίτον, ε, δράζεται στη ζήτηση. Δηλαδή ο όμιλος είναι ευέλικτο, αντιδρά και σε σχέση με τις ε, απαιτήσει αγοράς, αλλά και σε σχέση με ε, κρίσεις όπως είναι η COVID, η κλιματική αλλαγή κτλ. Και επίσης πολύ στενή συνεργασία με τις Εθνικές Τράπεζες Πρόθεσης για την αντιμετώπιση και των περιφερειακών αναγκών, των αναγκών της αγοράς, τα κράτη-μέλη και πάντα με βάση τις αρχές της προσθετικότητας και της επιλεξιμότητας. Έτσι εξυπηρετούνται περισσότερο οι χώρες ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητές τους. Και αυτό νομίζω είναι και μια πρόκληση για το μέλλον. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μόρτερ. Από ό,τι φαίνεται έχει συνδεθεί και μπορεί να μας μιλήσει ο κύριος Μακντάουελ. Παρακαλώ, κύριε Μακντάουελ, έχετε το λόγο. Mr. McDowell, please press the speak button. Thank you.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 Um, um, Παρακαλώ να περιοριστείτε στο δίλεπτο καθένας γιατί έχουμε μακροσκελή κατάλογο ομιλητών. Ξεκινάμε από τον κύριο Φερνάντες του ΕΛΚ. Yes. Can you hear me? are you? Μ' ακούτε? Θα προσπαθήσω να μιλήσω τα άσχημα αγγλικά μου. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο από το να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ για την οργάνωση της δημόσιας ακρόασης. Σε τομείς όπως ο τουρισμός και η υγεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα εργαλεία του. Έχουμε αρκετά μέσα να χρηματοδοτήσουμε τάχιστα την πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την ΕΤΕΠ και η χρηματοδότηση μικρών σχεδίων είναι δύσκολο έργο. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα πιο μικρά σχέδια, μικρή εμβέλεια σχέδια. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια είναι τα κονδύλια που έχει αφιερώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης από το COVID-19. Πώς μπορούμε να ανακάμψουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς μας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το InvestEU, το πρόγραμμα ε, για να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, ταχύτερα και καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Φερνάνδες. Η κυρία Περέιρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας και να θέσω κάποιε ερωτήσει στον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΠ, τον κύριο Μακδάουελ. Έχει τεράστια ευθύνη η ΕΤΕΠ για να στηρίξει την ανάκαμψη και να βοηθήσει κυρίω τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Τι τελευταίε εβδομάδε είχαμε ένα τεράστιο ασύμετρο, ε, συμμετρικό μάλλον υγειονομικό σοκ παντού, με αναπόφευκτες οικονομικέ συνέπειε, αλλά θα πρέπει και είναι καθήκον μα να μετριάσουμε την κρίση που θα έχει στο μέλλον ασύμετρα αποτελέσματα. Για να μην αφήσουμε λοιπόν καμία περιφέρεια πίσω, είτε στη φάση της ανάκαμψης λόγω έλλειψης ε, τεχνολογικών ή οικονομικών δυνατοτήτων να μοχλεύσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια με τον καλύτερο τρόπο και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα πρέπει ε, να βοηθήσουμε με κάποια κονδύλια από την ΕΤΕΠ, όπως έχουμε κάνει. Οι Εθνικές Αναπτυξιακές και Επιδετικές Τράπεζες θα έχουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αξιοποίησης ε, αυτών των κονδυλίων. Αλλά άλλη υποστήριξη αυτών, είναι διαφορετική υποστήριξη των τραπεζών αυτών στην Ευρώπη. Έχουμε ε, χώρες με διαφορετικές αναπτυξιακές και επενδυτικές τράπεζες, με πολύ πλούσια κεφάλαια δισεκατομμυρίων, ενώ άλλε χώρε έχουν μόνο μία επενδυτική τράπεζα με ελάχιστα κεφάλαια και χαμηλή επιχειρησιακή ικανότητα. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ λοιπόν. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να υπονομεύσει τι μικρομεσαίε των χωρών ε, αυτών που δεν έχουν ε, πλούσια παράδοση στις αναπτυξιακές ή επενδυτικές τράπεζες. Ή τι λύσεις μπορούμε να προσφέρουμε για να εξορροπήσουμε αυτές τις διαφορές. Έχω μία άλλη ερώτηση γιατί μια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι αναπτυξιακές ε, και επενδυτικές τράπεζες ε, θέλουν κυρίως να στηρίξουν την κεφαλαιοποίηση ε, των επιχειρήσεων αυτών στη φάση της ανάκαμψης. Ερωτώ λοιπόν, πώς μπορεί η ΕΤΕΠ να γίνει πλατφόρμα για να ενισχύσει τι διάφορε δομές και να βοηθήσει την κεφαλαιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τις εργασίες και δραστηριότητές τους στις πολυάριθμες ε, προκλήσεις ε, της, τεχνο... τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης ε, και τη ενεργειακή και περιβαλλοντική μετάβαση. Ευχαριστώ κυρία Περέρα. Ένα λουόμα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Καλημέρα σας από το Ελσίνκι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους καλεσμένους στο πάνελ για τις πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος αντιμετωπίζει πραγματικό οικονομικό σοκ και κραδασμούς που πλήττουν πολλές ε, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ως επακόλουθο του COVID-19. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε, να ενισχύσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αυτή την έκτακτη κρίση και να διαφυλάξουν τις θέσεις απασχόλησης. Χαίρομαι για τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ που ήταν σημαντικές μέχρι στιγμής. Ε, το Ταμείο Εγγυήσεων, το 25 δις, ένα άλλο μέτρο της ε, ΕΤΕΠ, είναι ευπρόσδεκτο βήμα, αλλά για να είναι αποτελεσματικό αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων θα πρέπει να συνδεθεί με την κρίση του COVID-19, ειδικά και να στηρίξει επενδύσει στην πραγματική οικονομία, στις πιο βιώσιμες επιχειρήσεις για να διαφυλάξουμε θέσεις απασχόλησης και όχι για να πληρώνουμε πρίμα των γενικών διευθυντών ή να καταβάλουμε μερίσματα. Επίσης, θα πρέπει η πολιτική μας αυτή να ευθυγραμμίζεται με τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, την πράσινη συμφωνία και τη δίκαιη μετάβαση. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε κυρίως αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνούμε και μια ανάγκη γεωγραφικής ισορροπίας στην κατανομή. Και να έχουμε υπόψη ότι οι τραπεζικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν μια πρόσθετη σημασία στις δραστηριότητες και να βοηθήσουν προσθέτω στις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Οπότε, ρωτώ την τράπεζα. Ε, πώς θα εξασφαλίσουν τη συμπερίληψη αυτών των κριτηρίων για την κατανομή και αποφύγουμε την ε, στήριξη μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Βέβαια, η κρίση δεν θα πρέπει να είναι πρόσχημα για την ε, άβληση των κριτηριών επιλογής. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί στην, στους όρους χρηματοδότησης για να υλοποιήσουμε στην, ε, την ανάκαμψη και να πιάσουν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων. Η δεύτερη ερώτησή μου ε, απευθύνεται στον κύριο Χαβιέρ Σόλ από τη μη κυβερνητική οργάνωση Counterbalance. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη η ΕΤΕΠ να επικαιροποιήσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και να συμπεριλάβει κάποια κοινωνικά κριτήρια και πτυχές. Γιατί οι δικαιούχοι σίγουρα δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Μάρκες για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για τις ε, εισηγήσεις. Οφείλω να σας πω ότι νιώθω κάποια απογοήτευση γιατί από τους εκπροσώπους της Τραπέζας Επενδύσεων και από τα Εθνικά Ταμεία Πρόθεσης συγκεκριμένα μέτρα ανταπόκριση και αντίδραση αυτή την κρίση. Και συνεχώς ακούμε πράγματα συνηθισμένα. Business as usual. Αυτά που λέγανε και χτες, τα λένε και τώρα, όμως για την σημερινή κρίση θέλουμε καινούργια πράγματα. Κάποια μέτρα που να μην είναι τα συνηθισμένα, τα τετριμένα. Και ερωτώ, του καλεσμένου μας και τον Αντιπρόεδρο. Πέστε μας τα εξαιρετικά μέτρα για να αντιδράσουμε σε αυτή την ε, κρίση. Το είπατε, Πρόεδρε, στην αρχή. Είχαμε εντυπωσιακή αύξηση των αποταμιεύσεων αυτό το δίμηνο. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή έπεσε εντυπωσιακά. Σταμάτησαν, φρέναραν οι επενδύσεις. Χρειαζόμαστε τώρα τις επενδύσεις, όχι στο μέλλον. Ε, διατέλεσα υπουργό στη χώρα μου και μπόρεσα μαζί με την ΕΤΕ να προωθήσουμε για τα νοικοκυριά την αποτελεσματικότητα της ενέργειας. Αλλά μου πήρε δύο χρόνια για να τα βρω με την ΕΤΕ. Μην πούμε πόσο πήρε για να έχουμε επιτόπου τις επενδύσεις να πιάνουν τόπο ας πούμε. Οπότε θα πρέπει τώρα κάτι να γίνει και όχι στο μέλλον. Πέστε μας ήδη τι έχετε εγκρίνει, τι μπορεί τώρα να γίνει μέτρα για μείωση επιτοκίων, αύξηση εγγύσεων, κινήσεις τώρα, κίνητρα. Κίνητρα που εγκρίθηκαν στο παρελθόν για να ενεργοποιηθούν τώρα. Τώρα θέλουμε κάτι το 20, ούτε το 21 ούτε το 22. Παρακαλώ να μου απαντήσετε αν μπορείτε, που ελπίζω. Ο πρόεδρος. Ο κύριος Μακντάουελ ε, βλέπουμε ότι συνδέθηκε οπότε να έχουμε τις υπόλοιπες ε, ερωταπαντήσεις και στη συνέχεια ο κύριος Μακντάουελ να μπορέσει τουλάχιστον να μας ε, μιλήσει σε σχέση με παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Οπότε, συνεχίζουμε. Μπίλι Kelleher για το Renew. Mr. Kelleher, please press the speak button. Thank you. Κύριε Kelleher, πατήστε το speak, το κουμπάκι που λέει speak. Mr. Kelleher, could you please... Κύριε Kelleher, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι. Yes. Hello. Ναι, ναι, μας ακούτε. Βλέπουμε μόνο το γραφείο του κυρίου Κέλεχερ όμως. Δεν βλέπουμε τον κύριο Κέλεχερ. Α, πρέπει να μετακινήσω την κάμερα. Λέει ο κύριος Κέλεχερ. Hello. We hear you, but we don't... Σας ακούμε, αλλά δεν σας βλέπουμε, λέει ο πρόεδρος. Είσαστε αλλού στο δωμάτιο. Τώρα θα πρέπει να είναι καλά, λέει ο κύριο Κέλεχερ. Οκ. Έτσι κι αλλιώ έχω ερωτήσεις να υποβάλω. Συμπαθάτε με. Ναι, ναι, πέστε μας, πέστε μας. Πρώτη ερώτηση. Προς τον κύριο Μακντάουαλ, τον αντιπρόεδρο. Όσον αφορά τον δανεισμό, τι προϋποθέσεις θα υπάρχουν από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, αλλά και από άλλους φορείς και έτσι να χορηγηθούν δάνεια σε ΜΜΕ. Να μην έχουμε δηλαδή κάτι σαν απλή υποκατάσταση στα συνήθη τραπεζικά δάνεια. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους δανεισμό μέσω των εθνικών τραπεζών αλλά όχι επιπλέον πόρους. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πραγματική οικονομία παίρνει παραπάνω πόρους. Μην έχουμε απλώς υποκατάσταση αυτών που ήδη θα, έτσι κι αλλιώς θα δανείζονται από τις τράπεζες. Επίσης, όταν οι τράπεζες αξιολογούν το αξιόχρεο των οφηλετών, τι προϋποθέσεις και κριτήρια εσείς θα θεσπίσετε για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει δίκαιη αξιολόγηση, αντικειμενική, αμερόληπτη και ότι οι τράπεζες δεν αμείβουν, δεν ε, αβαντάρουν τους καλούς τους πελάτες ότι θα πρέπει να αξιολογούνται τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά μόνο. Τελικά, πες μας θα υπάρξει κάποιος επιτητητής ο οποίος να αξιολογήσει κάποια δάνεια τα οποία έχουν απορριφθεί ως αιτήσει. Αυτές οι τρεις ερωτήσεις από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα έχουμε τον κύριο Χώσικ, ο οποίος επίσης αντιπροσωπεύει το Renew. Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ έχω ρωτήσει προς τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕ. Γιατί νομίζω ότι οι πόροι κυρίως από εκεί θα προέλθουν για την υπόθεση της ανάκαμψης μεσογητής για τα σχετικά με την ΕΤΕ. Βρίσκαστε σε φάση θετικής μετάβασης. Καλά τα πάτε και συνεχίστε. Όσον αφορά την προσπάθεια για το κλίμα, ενώ Σλοβακία και Τσεχία έχουμε μία χωρίς προηγούμενο ξηρασία. Και τι γίνεται με την πράσινη αιρεσιμότητα. Συνεχώς συζητείται η υπόθεση των περιβαλλοντικών επενδύσεων σε σχετικά έργα κλπ. Αλλά το σημαντικό είναι να υπάρχει συνοχή στην πολιτική. Να γιατί έχει σημασία η αιρεσιμότητα. Οπότε τα επενδυόμουν από την ΕΤΕ να βοηθούν και να μην δυναμητίζουν αυτή την προσπάθεια. Η ΕΤΕ συμμετέχει στην τεχνική ομάδα για αυτό που λέμε ταξόνομη. Άρα, εσείς τι θα κάνετε όσον αφορά την πολιτική των επιχορηγήσεων και δανεισμού πρόκειται να διατεθούν για την ανάκαμψη πολύ σημαντικοί πόροι. Άρα εσείς πώς θα υποπτεύσετε. Και επίσης πώς θα εφαρμόσετε το μέτρο διευκόλυνσης χρηματοδότησης κεφαλαίου. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. και για τα δάση και γενικότερα για την περιβαλλοντική πολιτική που έχει σχέση με τη βιοπικιλότητα. Και έτσι θα δοθούν και ευκαιρίες στην απασχόληση. Τέλος. Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, εδώ αναδείπτει κάποιες ευκαιρίες. για τα απόβλητα, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για τη μεταφορά τεχνολογίας. Οπότε έτσι υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης ΜΜΕ και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία των ΜΜΕ ενώ ταυτόχρονα βοηθούνται ή βοηθάται τέλο πάντων η, η επίτευξη των στόχων του περιβάλλοντος. Προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να σας δούμε να κινήσετε. Ο Πρόεδρος. Ντονάτο. ID. Mrs. Donato, could you press the... Κυρία Ντονάτο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι που λέει speak. Εδώ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Με ακούτε, λέει η κυρία Ντονάτο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ε, ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές για τα όσα είπανε στην ακρόαση ε, βέβαια και τους ευχαριστώ για τις προσπάθειες που γίνονται. Ε, είναι προς, συνεχής οι προσπάθειές σας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της υποστήριξης, δηλαδή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Δυστυχώς όμως, Ακριβώς όπως είπαν και οι συνάδελφοι που προλάλησαν, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν τα πάμε καλά όσον αφορά στην ε, αλυσίδα, στη διαδοχή για την δανειοδότηση. Αυτά και στη δική μου περιφέρεια, το νότο της Ιταλίας, δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει ε, μια τέτοια, μια τέτοια προβληματική κατάσταση για τη χορήγηση των δανείων στις ΜΜΕ και έχουμε κάποιες καθυστερήσεις σε αυτή τη χορήγηση γιατί τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν έχουν σχέση με την ε, ανακύκλωση, αλλά επίσης και θέματα σχετικά με το πτωχευτικό δίκαιο. Ε, και τελικά οι τράπεζες όπως ε, διαπιστώθηκε έχουν κάποιο είδους ε, ασυλία, ποινική ασυλία. Οπότε θα πρέπει η να κινηθεί πάνω από αυτό το κατόφλι των 2 εκατομμυρίων. Όμως αυτό δεν προβλέπεται για τον προ καταρκτικό σχεδιασμό αυτής της χρηματοδότησης. Επομένως, δεν θα πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα όσον αφορά τους ΟΤΑ στη δική μας περιφέρεια. Γιατί έχουμε κάποια μικρότερα προγράμματα και έργα ε, και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά οι πιο φτωχοί ΟΤΑ. Οπότε χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη προσπάθεια όσον αφορά τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επιχειρήσεις, ε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις κρατικές αρχές σε μας στο Νότο και θα πρέπει έτσι να αξιοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερο αυτές οι παρεχόμενες δυνατότητες και οι ενέργειες της ΕΤΕΝ να πιάσουν ε, τόπο και να βελτιωθούν αυτοί στους οποίους στοχεύουν αυτά τα μέτρα. Thank I now go to Madam Bonfrisco uh, ID. Bonfrisco ID. Grazie. Σας ευχαριστώ, λέει κυρία Μπονφρίσκο. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ε, ευκαιρία να μιλήσουμε και να μιλήσουμε αυτούς τους σημαντικούς καλμένους. Έχω δύο ερωτήσεις για τον αντιπρόεδρο της ΜΠΕ. Σε αυτά τα κριτήρια της ε, αξιολόγησης ε, σήμερα θέλουμε να δούμε το πώς η ισορροπία των ε, κρατών μελών στις κρατικές επιχορηγήσεις καλύπτει και το ότι υπάρχει μια μεγάλη ανισορροπία σε σχέση με την Γερμανία. Η ΕΤΕ μπορεί και αυτό να το μετρήσει όσον αφορά την εκταμείευση της χρηματοδότησης. Δεύτερος για τον κύριο ε, Παλέρμο. Το ταμείο σας τι εμπειρία έχει αποκτήσει όσον αφορά τη βοήθεια, τη χρηματοδότηση του πλάνου Juncker. Στήριξε τη χώρα μας σημαντικά όσον αφορά τα θέματα της ψηφιακής υποδομής. Και μια τελευταία ερώτηση. Για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και για το τι γίνεται με τους ε, φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν και στην Ευρώπη σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα από ποτέ. Θα πρέπει να προσέξουμε οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕ να μην βοηθήσουν κάποιες δραστηριότητε, οι οποίες στη συνέχεια θα φέρουν ε, μια διάλυση του οικονομικού ιστού των κρατών μελών. Thank you very much. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Τον ξαναχάσαμε τον κύριο Μακντάουελ, από ό,τι φαίνεται ή όχι. Όχι, δεν τον χάσαμε, τον έχουμε τον κύριο Μακντάουελ. Αν με ακούτε κύριε Μακντάουελ, θα ήθελα να σας δώσω τώρα το λόγο. Φαντάζομαι ότι ακούσατε τις παρεμβάσεις, ακούσατε τις ερωτήσεις ε, των Ευρωβουλευτών και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εστιάσετε στις απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις ε, για τα επόμενα λεπτά. Έχετε παρακαλώ το λόγο. Are Τον χάσαμε. Τον αντιπρόεδρο. Ο κύριος Μόλτερ λοιπόν ίσως θα μπορέσει στη θέση του κύριου Μακντάλ να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν και αφορούσαν το ΕΦΣΥ. Κύριε Μόλτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω το εξής, γιατί κάποιοι μίλησαν για τη διακυβέρνηση και για την ικανότητα επιτέλους του έργου μας επιτόπου σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ. Θέλω να επαναλάβω λοιπόν τις παρατηρήσεις που έκανα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Κόμβο, το Advisory Hub. Θεωρώ ότι το συμβουλευτικό σκέλος είναι το, ένα από τα πιο σημαντικά και για τον ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους φορείς. Αυτό το hub θα πρέπει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στη μελλοντική προοπτική του InvestEU. Δεύτερον, η συνεργασία με τις εθνικές τράπεζες ή οργανισμούς πρόθεσης είναι ένας τρόπος πολύ θεμελιώδης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα αλλά και συνυπολογισμό των αναγκών της αγοράς που είναι τελείως διαφορετικές σε κάθε χώρα. Και όπως είπε και ένας συνάδελφός σας, αν δεν υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο σε όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που έχουν αυτοί οι θεσμοί, ε, πρέπει να το έχουμε υπόψη, διότι οι επενδύσει σε αυτόν τον τομέα θα αυξήσουν την αξία εξορισμού και ο κόμβος, ο συμβουλευτικός, έχει το ρόλο του γιατί ακριβώς παρέχει στοιχεία για να βοηθηθούν αυτοί οι φόρεις. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για το τρίτο στοιχείο που είναι οι επενδυτικές πλατφόρμες που προβλέπονταν ως ε, ένας μηχανισμός δημιουργίας αποτελεσμάτων όταν ε, εμείς και το είδαμε και με το CTP, το ιταλικό. Έχουμε και για τις πλατφόρμες και για, το, για την πλατφόρμα, για το παράθυρο καινοτομία κάποιες πλατφόρμες ε, για να έχουν ένα ρόλο και στο μέλλον και στο πλαίσιο του InvestEU. Έχουμε τέσσερις για το ΕΦΣΙ και δύο για το παράθυρο καινοτομία, τέτοιε πλατφόρμες. Επίσης, να σας πω ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε ήδη από τώρα ε, μελλοντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, το ΕΟ, ε, ε, InvestEU κτλ. Και θα πρέπει να έχουμε τις επιχορηγήσεις από διαδροτικά ταμεία ή το Ταμείο γεωργικής Ανάπτυξης. Πρέπει να συνδυάσουμε ΕΦΣΙ και ΕΣΥΦ. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τη μελλοντική προοπτική. Δηλαδή, ταμείο στρατικών επενδύσεων και επενδυτικά ταμεία. Επειδή πολλοί μίλησαν για την ανταπόκριση στην κρίση, για την ανταπόκριση στην COVID-19, πρέπει να σας πω ότι βεβαίως και περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ό,τι αφορά το ΠΔΠ για τα επόμενα έτη, για το 2021 και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά περιμένουμε επίσης και την επαναδιατύπωση του InvestEU, τον επανασχεδιασμό. Έχουμε δε και το Solvency το πρόγραμμα που πρέπει ε, επίσης να ε, έχουμε την πρόταση, τη σχετική. Και μάλλον αύριο θα έχουμε ε, μια πρόταση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδώσει. Για το ETF περί αυτού πρόκειται επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά μακάρι να μπορέσει ο κ. Μακντάουλ, αντιπρόεδρο. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύσεων. Καλό θα ήταν να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το ταμείο. Και τέλος, σίγουρα έχουμε τον τομέα της υγείας και τον τομέα του τουρισμού. Ιδίω στο πλαίσιο του παραθύρου των ΜΜΕ. Έχουμε εστιάσει αυτούς τους τομείς που είναι οι πλέον πληγέντες το ΕΦΣΙ, το InvestEU, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα μέτω στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου νομίζω θα πρέπει να εστιάσουν πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα και να παράσχουν άμεση ε, πραγματική υποστήριξη, γρήγορη υποστήριξη σε αυτούς τους τομείς. Και αυτό δεν είναι σε αντίφαση με το πράσινο οικονομία, στόχο για την αλλαγή του κλίματος. Πρέπει να ε, μείνουμε σε καλή τροχιά, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε να είναι ανθεκτική ένωση, ε, γιατί αυτό μετράει. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μόλτερερ. Ο κύριος Παλέρμο ε, θα πάρει τώρα το λόγο γιατί και αυτός ήταν ε, νομίζω αποδέκτης κάποιων ερωτήσεων. Κύριε Παλέμο, έχετε το λόγο. Ε, thank you. Σας ευχαριστώ. Η τράπεζά μας αντέδρασε άμεσα στην πανδημία COVID θεσπίζοντας από κοινού με την Ιταλική κυβέρνηση κοινά μέτρα. Έχουμε εξασφαλίσει αρκετή ρευστότητα στο σύστημα με πολλά μέτρα που άμεσα και έμεσα χρησιμοποίησαν το τραπεζικό σύστημα για να εξασφαλιστεί ρευστότητα σε όλους τους τομείς που επηρεάστηκαν και επλήγησαν από την COVID-19. Επίσης, από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε προσφέρει και εγγύσεις ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν άμεσα τους, τον τους τομείς που έχουν πληγεί με πάνω από 100 εκατομμύρια εγγύσεων. Επίσης, στηρίζουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με άμεσες επενδύσεις αυτές και ήδη τα μέτρα αυτά έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Όμιλο ΕΤΕΠ, πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως αυτές του κόσμου, του προγράμματο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μια άλλη πρωτοβουλία που ε, ανέλαβε η ΕΤΕΠ είναι πρόγραμμα COVID με εγγύηση ύψους 200 δις. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα να επικεντρωθεί κυρίως σε τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερως από την κρίση COVID. Και τομείς κυρίως όπως ο τουρισμός και η συναφής με αυτόν κλάδι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες ερωτήσεις. Το επενδυτικό σχέδιο Juncker ε, στέφθη με μεγάλη επιτυχία κατά τη γνώμη μας. Έχουμε επενδυτικές πλατφόρμες με 4 δις και ένα μεγάλο τμήμα ήδη έχει εκταμιευτεί. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε άμεσα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες και όλες οι πρωτοβουλίες μας αυτή την άγουσα ακολουθούν. Ε, και επίσης παρακολουθούμε και τον αντίκτυπο των επενδύσεων μας. Όπως ξέρετε αυτή η κρίση είναι ιδιάζουσα. Μεταξύ άλλων και για το λόγο ότι Τα περισσότερα, οι περισσότεροι οργανισμοί προσπαθούν να εργαστούν όλο πιο, πιο έξυπνα και αποτελεσματικά, κάτι που θα πρέπει να στηριχθεί στις επιμέρους χώρες. Οπότε θα πρέπει να απλουστεύσουμε την διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα της οικονομίας τους σπόρους γιατί επαναλαμβάνω η κρίση αυτή είναι ιδιόμορφη και πρωτοφανής γιατί όλο και περισσότεροι εργάζονται από το σπίτι, έχουμε τηλεργασία, κάτι που καθιστά πιο ε, περίπλοκη ακόμη τη διαχείριση της συγκεκριμένη κρίσης. Ευχαριστώ κύριε Παλέρμο. Κύριε Σόλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Στην ερώτηση του κυρίου ελουόμα, θα ήθελα να πω ότι σίγουρα πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη ε, η ΕΤΕ να αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο των σχεδίων που χρηματοδοτεί. Επίσης, να αναθεωρήσει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά της πρότυπα. Θα ξεκινήσει η σχετική επανεξέταση στα τέλη του 2020, να ληφθεί καλύτερα υπόψη η συνοχή, η κοινωνική συνοχή, στον τρόπο επιλογή και αξιολόγηση των σχεδίων. Θα πρέπει και οι κοινωνικέ ανισότητε να συμπεριληφθούν ω κριτήριο και ο αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα των σχεδίων που χρηματοδοτούνται ή στηρίζονται από την ΕΤΕΠ. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, το 2019 η ΕΤΕΠ πέρυσι υιοθέτησε μια νέα πολιτική για τη φορολογία που βελτιώνει την προηγούμενη της πολιτική. Υπάρχουν όμως κάποια εκκρεμή θέματα ακόμη. Για παράδειγμα, η ΕΤΕΠ δεν απαιτεί από τους πελάτες της να, κάνουν, να υποβάλουν εκθέσεις χώρα. Οπότε θα δούμε πώς η νέα φορολογική πολιτική της ΕΤΕΠ θα εφαρμοστεί εμπράκτο και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Ε, να δίνονται αναφορές και να λογοδοτεί η ΕΤΕΠ ε, στο Κοινοβούλιο και να ενημερώνει και τον κόσμο πώς εμπράκτως εφαρμόζεται η νέα φορολογική της πολιτική. Και επανέρχομαι στο θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ΕΤΕΠ δεν ε, χρηματοδοτεί άμεσα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, περνά από ενδιάμεσου χρηματοοικονομικούς οργανισμού και κυρίω από ε, εμπορικέ τράπεζε που δίνουν πιστοτικέ ε, γραμμέ και κονδύλια και δάνεια. Εδώ θα πρέπει να εμείνουμε ιδιαίτερα στην ανάγκη διαφάνεια αυτών των δραστηριοτήτων. Όταν χρησιμοποιεί κάποιο ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού οργανισμού, θα πρέπει να κρατά τον έλεγχο για το πού πηγαίνουν, πού καταλήγουν τα δημόσια κονδύλια. Και θα πρέπει να γίνεται τέτοιο έλεγχο όπω και στα άμεσα δάνεια. Και υπάρχει και το θέμα τη προσθετικότητα. Πώ αυτά τα κονδύλια, πώ αυτά τα δάνεια θα ε, επιτρέψει οι τράπεζε να κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν διαφορετικά. Και εδώ ε, θα παίξει κάποιο ρόλο το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στην δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να είναι προσθετική αυτή η ενίσχυση. Και κάθε δημόσια τράπεζα ενδιαφέρεται, αλλά θα πρέπει ο κοινοτικό προπολογισμό να έχει πραγματικά ένα προσθετικό, συμπληρωματικό αποτέλεσμα. Και θα ολοκληρώσουμε το θέμα του βραχυπρόθεσμου αντικτύπου και της υποστήριξης. Ο, σχέδιο, ο κύκλος των σχεδίων είναι αρκετά μακροπρόθεσμος στην ΕΤΕΠ για εύλογους και ευνόητους λόγους. Χρειάζεται μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση των σχεδίων. Οπότε υπάρχουν κάποια όρια στις δραστηριότητες, βραχυπρόθεσμε βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες της τράπεζας. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ μιας μακροπρόθεσμη προοπτική στις δραστηριότητες τη ΕΤΕΠ, σε συνδυασμό και με την Πράσινη Συμφωνία και με πιο μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επενδύσει στην ενεργειακή απόδοση, στην καινοτομία, στην αποκέντρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, επενδύσει στην κυκλική οικονομία. Αυτό ήταν ένα καλό δρόμο για να ακολουθήσει το μέλλον η ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ. Δυστυχώ δεν έχουμε ακόμη επαφή με τον κύριο Μακτάουελ, οπότε θα ζητήσουμε να απαντήσει γραπτό το συντομότερο δυνατό σε ερωτήσει. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερα μπορούμε να κάνουμε δεδομένων των συνθήκων. Τώρα για το δεύτερο τμήμα. Και τώρα να δώσω. Θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο τη ΕΚΟΝ. Δώσω το λόγο στην. Ε, Σε ευχαριστώ, Συμπρόεδρε. Τώρα αρχίζει ο τρίτο ε, γύρο των ερώτων απαντήσεων για να δώσουμε τον λόγο πρώτα απ' στον David Κόρμαντ της Επιτροπής των Προϋπολογισμών που προέρχεται από τους Πράσινους. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω με ακούτε και σας ευχαριστώ για τα όσα μας εξηγήσατε. Μπράβο για αυτήν την ε, συνάντηση. Ε, βέβαια, γίνεται σημαντικός ο ρόλος σας όσον αφορά την ανάκαμψη και το μέλλον της Ευρώπης, αλλά δεν ακούγεται καθόλου καλά ο κύριος Κορμά. Θα πρέπει να βρεθούν τα μέσα για τωρινή αντίδραση στην κρίση αλλά και για το μέλλον, για τις ΜΜΕ και ευρύτερα και πριν την κρίση της πανδημίας. Λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνει τράπεζα για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και το βέβαιο είναι ότι με αυτή την ε, πανδημία, ε, αυτή η φιλοδοξία δεν θα πρέπει να μπει στο χρονοτούλαπο. Οπότε, θα πρέπει να συνδέσουμε την περιβαλλοντική κρίση με την υγειονομική κρίση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στις χρηματοδοτήσεις. Διακόπτε το κύριο Σαρμό. ακούγεται ο κύριος Κορμό. Έχει διακοπή σύνδεση με τον κύριο Κορμό. Κυρία Πρόεδρε, δώστε το λόγο αν θέλετε στον επόμενο μιλήτη. Κυρία Τινάλη, δυστυχώ. Όλα εξαρτώνται από την συσκευή που έχει ο καθένα. Οπότε πάμε τώρα στον επόμενο που είναι ο Μπάσικ Χάουτ τη Οικονομική Επιτροπή και αυτό πράσινο. Ο κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ελπίζω ότι η δική μου σύνδεση θα είναι πιο σταθερή. Είχα κάποιε ερωτήσεις ε, που έχουν σχέση με αυτά που έλεγε ο κύριος Κορμό, οπότε είναι σημαντικό να τον ακούσουμε. Τέλος πάντων, η ερωτήση είναι προς τον κύριο Μακντάουλ. Ε, όταν έχουμε ακρόαση με την ΕΤΕ, βέβαια, Κρίμα να μην έχουμε κάποιον από την ΕΤΕ για να μας τα πει, για να μας απαντήσει. Οπότε όλα αυτά είναι κάπως ε, αδέξια, να πω το το. Ελπίζω ότι τουλάχιστον ως κύριος Μακντάουλ και εγώ θέλω να προσέξουμε το θέμα του Ταμείου Εγγύσεων για την πανδημία. Αύριο θα δημοσιοποιηθούν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε θα έχουμε και τον πυλώνα του InvestEU Οπότε θα είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάληψη πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και ελπίζω σύντομα να μας τα απαντήσει αυτά όλα τα ερωτήματα γιατί κατεπήγουν ο κύριος Μακντάβελ. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κλιματική κρίση και ο κύριος Αρμόν εκεί ε, το πήγαινε. Αλλά θα ήθελα να είναι πιο ξεκάθαρη η ΕΤΕ γιατί αν κοιτάξουμε το website και διαβάσουμε τι λέει για το Ταμείο Εγγύησης λέει ότι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ουσιαστικά τις επενδύσεις για την ανάκαψη στην Ευρώπη μόλις περάσουν τα χειρότερα τα σχετικά με την πανδημία. Εμένα μου φαίνεται κάπως περίεργη αυτή η διατύπωση γιατί πώς θα κρυθεί το πότε πέρασαν τα χειρότερα τι εννοείται, γιατί νομίζω ότι η οικονομική κρίση που έρχεται αυτή θα είναι τα χειρότερα. Δεν τα έχουμε δει τα χειρότερα ακόμα. Και τι λέει η ΕΤΕ, ότι ναι, πρέπει να το συνδέσουμε το θέμα και με την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει πιο ξεκάθαρα να εξηγήσει η ΕΤΕ τι εννοεί με αυτήν την διατύπωση και πιο συγκεκριμένα πότε θεωρείται θα πρέπει να έχουμε ε, μια πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα με την ιδιότητά της ως κλιματικής τράπεζας. Δεν λέει τίποτα επομένω η εν λόγω φράση στο website. Τώρα κάτι άλλο για την ισότητα των όρων. Το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι. Αν δούμε τι γίνεται για τις κρατικές ενισχύσεις, έχουμε πάνω από δύο τρεις, τα μισά γερμανικά. Οπότε δεν αυτό δεν είναι και πολύ ισότητα όρων του ανταγωνισμού για την αγορά και τα πράγματα γίνονται χειρότερα από τις κρατικές επιχορηγήσεις ε, και το πράσινο φως που έχει δώσει για αυτές τις επιχορηγήσεις, για φέτος η Κομισιόν, άρα κερδισμένε είναι μόνο ισχυρέ χώρες. Για κοιτάξτε από πλευρά Ένωση, ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει αυτοί που έχουν λιγότερα φορολογικά έσοδα να, και δημοσιονομικά να βοηθηθούν. Τι θα κάνει το Ταμείο Εγγύσεων, πώς θα εξασφαλίσουμε το ότι όταν προχωρήσουμε με το Invest EU ε, θα βοηθήσει και το Invest EU. Τα είπε ο κ. Μόλτικερ. Τι θα κάνει το ΕΦΣΕ. Πέστε μας όμως συγκεκριμένα Διαβεβαιώστε μας ότι θα το φροντίσετε το πρόβλημα, αλλιώ δεν θα τα πάμε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Μπάς και... Α, να, ο, ο κύριος Κορμόν τώρα έχει καλύτερη σύνδεση. Και πάλι κοντά μας. Για να δούμε. Έχετε το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Α, Ούτε τώρα έχει καλή σύνδεση ο κύριος Κορμού. Όχι, όχι, κόπηκε πάλι η σύνδεση του κύριου Κορμού. Yes, apparently. Ναι, ναι. Η σύνδεση με τον Νταβίδ δεν είναι σταθερή. Αλλά ο κύριος Μακντάουλ είπε ότι θα απαντήσει εγγράφο γιατί ούτε αυτός μπορεί να συνδεθεί καλά. Άρα, να μας υποβάλει τις ερωτήσεις του ο κύριος ε, Κορμό, να υποβάλει τις ερωτήσεις τον κύριο Μακντάουλ και να του απαντήσει οπότε όλοι, όλοι, όλοι να καλυφθούν. Και τώρα ο κύριος Μπόγκταν Ζόγκα για το ECR, Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εγώ τώρα θέλω να επανέλθω σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι το θέμα της ε, υγείας. Πρόκειται για μια πανδημία η οποία είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις και γι' αυτό και σας ε, ερωτώ και θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Οι εθνικές... Είναι πραγματικά πρωτοφανής αυτή η κατάσταση η υγεία των πολιτών απειλείται, τα κράτη μερικές φορές είναι ανήμπορα και μερικές φορές γίνεται και πραγματικά μια βάναυση επιλογή των αρρώστων, ε, ε, μερικών που δικαιούνται ε, θεραπείες και άλλων για τους οποίους δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα ή μέσα. Πότε ε, πιστεύετε θα πρέπει να δράσουμε και να παρεύουμε και σε αυτό το τομέα και να βοηθήσουμε τις δημόσιες διοικήσεις, τις εθνικές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί έτσι θα εξορροπήσουμε ε, τις ανισότητες. Είτε με εγγύησεις χρηματοδοτικές, είτε με χρηματοδότηση του τομέα της υγείας. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των πολιτών. Δεύτερη ερώτηση. Ε, σίγουρα η πανδημία κλώνησε και την υγεία, κλώνησε την οικονομία, ίσως κλώνησε και άλλους τομείς, όπως την ενέργεια. Ίσως η ΕΤΕΠ ε, θα, θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη σε ό,τι αφορά τη μη χρηματοδότηση κάποιων ε, επενδύσεων χαμηλών εκπομπών στο φυσικό αέριο. Για να μην έχουμε κάποια προσδόκητα δράματα και τραγωδίες στο μέλλον από την πλευρά αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τους δύο τελευταίους ομιλητές από την ΚΟΕ, Κρίς Μακμάνος. Mr. McManus, please press the speak button. Thank you. Παρακαλώ πατήστε το κουμπί κύριε Μακμάνος. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους πανελίστες. Και ελπίζω ο συμπατριώτης μου ο κύριος Μακδάρ τουλάχιστον να ακούει τα σχόλιά μου. Νιώθουμε μεγάλη απογοήτευση. Έχουμε την ΕΤΕΠ, ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που θα επενδύσει υποτίθεται στις υποδομές ε, και θα έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα για να τονώσει και την οικονομία. Ε, οπότε, αντί να χρησιμοποιούμε τον όμιλο ΕΤΕΠ ε, για την ανάκαμψη, ίσως θα πρέπει να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, συνδυάσει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το α, σχέδιο για την ανάκαμψη. Και νομίζω ότι έχει πιστεί και ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε όμως περιορισμένο ε, προϋπολογισμό στην ΚΑΠ, για παράδειγμα, και θα ήθελα εκεί η ΕΤΕΠ ε, να παίξει κεντρικό ρόλο, πρωταγωνιστικό και όχι παρεμπίπτοντα και περιθωριακό. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι οι ανώτατες νομικές ικανότητες ε, της ΕΤΕΠ που θα μπορούσαν και θα όφυλα να χρησιμοποιήσουν και γιατί δεν είναι πρωταγωνίστρια ΕΤΕΠ και ε, να μην έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέε εξουσίε. Δεν θα πρέπει η ΕΤΕΠ να υπενθυμίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλου ότι υπάρχει και ότι θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Επίση, θα πρέπει όλοι οι δικαιούχοι να πληρούν όχι μόνο του περιβαλλοντικού αλλά και του κοινωνικού στόχου. Και να μην χρηματοδοτείται καμία επιχείρηση που απολύει ε, εργαζόμενους ή καταβάλει μερίσματα. Πώς μπορεί το Κοινοβούλιο και η ΕΤΕΠ να καταστήσουν αυτές τις προϋποθέσεις στον κανόνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Πέτρος Κόκαλης τώρα από την ΚΟΕ. Hello and uh, thank you for this conversation. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Είμαι ο τελευταίος ομιλητής, έχω μια γενική παρατήρηση. Θα ήθελα να συγχαρώ την ΕΤΕΠ για τον οδικό χάρτη για το κλίμα, μια και θα μετατραπεί σε τράπεζα για το κλίμα, και χρήση του 50% ε, του συνολικού κονδυλίου για το κλίμα και το άλλο 50% που θα πρέπει να πληρεί την αρχή του μη βλάπτη και ε, χρήση της ταξινομίας, φαντάζομαι δεν αρκεί να έχουμε μισή ε, ρυθμίση για το κλίμα. Θέλουμε ολοκληρωτική. Επίσης, πιστεύετε ότι τα αντισταθμίσματα της βιο ποικιλότητα και το αντιστάθμισμα του άνθρακα αρκούν για να προστατεύσουν τη φύση. Επίσης, μιλήστε για τις ε, πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας ε, για την καινοτομία. Μπορείτε να μας ενημερώσετε περαιτέρω. Χθες είχαμε μία επιστολή 8 χωρών μελών που ζήτησαν εξαιρέσεις από την απαγόρευση της χρηματοδότησης των ορυκτών καυσίμων. Πιστεύετε ότι τα ορυκτά καύσιμα θα μπορούσαν να γίνουν μια γέφυρα, ένα μεταβατικό στάδιο για να υλοποιήσουμε την κλιματική ουδετερότητα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πατήστε κυρία Πρόεδρε το κουμπί speak. Α, με συγχωρείτε, ευχαριστώ. Κυρία Τινάλη, με αυτή την ε, Τελευταία ερώτηση. Θα περάσουμε ε, στις απαντήσεις από τους ε, ομιλητές μας. Και όπως προείπα θα απαντήσει γραπτός ο κύριος Μακντάουελ. Με αυτή λοιπόν ε, την προϋπόθεση δίνω το λόγο ξανά στον κύριο Μόλτερερ. ο οποίος κόβεται. Sorry, I think now it is... Συγγνώμη, τώρα λέει δουλεύει το σύστημα. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Να σας διαβεβαιώσω θα μιλήσω με τον Άντρου Μακντάουελ και θα το μεταφέρω και την ουσία αλλά και τον τόνο, το ύφος των ερωτήσεων ώστε να μπορέσει να απαντήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν μου επιτρέπετε δύο λόγια για αυτό το ευρωπαϊκό και αυτή την ευρωπαϊκή πανευρωπαϊκή εγγύηση που βασίζεται 25 δις από τις ε, χώρες ε, που θα μοχλεύσει πολλά δις ε, και μάλλον αναμένουμε σύντομα να μπορέσει να δρομολογηθεί, γιατί τα κράτη-μέλη δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Ε, δεν είναι λοιπόν σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα στηρίξει το ποσό αυτών και των 250 που θα μοχλευτούν θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αντιμετωπίσει την κρίση και θα βοηθήσει και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανταπόκρισης ε, στην πανδημία. Αυτό εφόσον και αγκριθεί αμέσως, εφόσον αγκριθεί από το ΔΣ Περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν αύριο, το είπατε και μερικοί από εσά και αυτό θα επηρεάσει και τη δράση της ΕΤΕΠ από φέτο. Εφόσον προβλέπετε ότι το ΕΦΣΥ θα έχει ένα νέο παράθυρο, Solvency Window, το οποίο ήδη από φέτο είναι έτοιμο και θα περάσει στο InvestEU. Μαζί με άλλες δυνατότητε για του χρόνου. Μια παρατήρηση για τον Μπάς. Μην βασίζεσαι τόσο στο χρώμα των ματιών, αλλά στα γεγονότα που μιλάνε από μόνα τους. Από τότε που ξεκινήσαμε το ε, ταξίδι μας, ε, έχουμε καλύψει όλα τα κρατημέλη. Υπήρξε μια φάση ε, που έπρεπε να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος τα νεα αυτά τα οποία είχαν πληγεί από την κρίση, τα νότια κράτη αυτό που είπε ε, και ο Έλληνας συνάδελφος ε, και το CDP είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες ε, και οι δευτερότητες των περιοχών. Και αυτό θα γίνει και στο InvestEU, που γι' αυτό έχει τώρα αυτό 75% εγγύηση από την ΕΤΕΠ και 25% από εθνικές τράπεζες και οργανισμούς προώθησης. Αλλά, για να το πω και πιο ομά, από εμά θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξει ετοιμότητα και πολιτική υποστήριξη από τις κυβερνήσει των κρατών μελών για να ενισχυθούν οι ε, φορεί αυτοί. Το CTP είναι ένα παράδειγμα που πραγματικά ε, δείχνουμε ότι πώ όταν ε, το κράτος στηρίζει, το Ιταλικό στην προκειμένη περίπτωση, μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένα πράγματα με πολύ καλό τρόπο. Κύριε Κάουτα, Είπατε τι άλλε ιδέε υπάρχουν. Είπα, οι επενδυτικέ πλατφόρμε μπορούν να διαδραματίσουν έναν περισσότερο ε, ρόλο. σω μέσω και του κανονισμού InvestEU θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα. Δεν με ικανοποιεί τόσο πολύ το τι θα γίνει με τα διαρθρωτικά ταμεία και το ESIF και πώς θα συνδυαστεί με το EFSI και αργότερα με το InvestEU το Omnibus βοηθούσε, αλλά δεν βελτίωσε πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι νομικό το ζήτημα. Ε, πρέπει και οι εθνικές τράπεζες και φορείς πρόθεσης και τα εργαλεία όπως οι πλατφόρμες ή το blending αυτό, EFSI και ΕΣΥΦ. Αυτό είναι που θα βοηθήσει για να βοηθήσουμε τη συνοχή και τη δίκαιη κατανομή, το δίκαιο επιμερισμό. Και αυτό να ισχύει για το μέλλον. Η εμπειρία του EFSI... Ε, δείχνει ότι ναι, κάναμε πρόοδο, όμως περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και σας είπα και κάποιες ιδέες μόλις τώρα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παλέρμο, εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε. Νομίζω ότι πράγματι έχουν τους τελευταίους μήνες τέθη σε εφαρμογή πολλά ε, μέτρα και εργαλεία και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ σας είπα για την Ιταλία. Νομίζω ότι τώρα το θέμα είναι να αντιδράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο, να έχουμε αυτή τη ρευστότητα, αυτές τις εγγύσεις, τη στήριξη αυτή, την κεφαλαιακή, για όλους τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο. Η Ευρώπη νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξει τους τομείς που ανοίγουν ευκαιρίες για μελλοντική πρόοδο. Όχι να στηρίξει μόνο τις μεγάλες εταιρείες, αλλά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Που πολλές φορές βρίσκονται και πίσω από τις μεγαλύτερες τομές μηχανολογίας, ενέργειας, δίκτυα, υγεία, τουρισμός, μεταφορές είναι τομείς νευραλγικοί και θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες προσεχείς μήνες. Δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε τις δυσκολίες αυτές αυτή τη στιγμή, άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλοι οι εθνικοί φορείς και η ΕΤΕΠ θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να αντιδράσουν και να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα εφόσον αυτά χρειαστούν ή να τα προσαρμόσουν ώστε να είναι πλέον αποτελεσματικά. τέλει, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, νομίζω ότι για το μέλλον θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για ενεργειακή μετάβαση το CDP εστιάζει στη βιωσιμότητα, στην αηφορία. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Και πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα, η αηφορία είναι ένας τομέας που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη όλης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο μέλλον. Και να βοηθήσει πολλούς και διάφορους τομείς στην Ευρώπη. Να είναι ο μοχλός της μελλοντικής ανάπτυξης Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χαβιέρ Σόλ τώρα. Πατήστε το κουμπί, κύριε Σόλ. Ευχαριστώ σε ό,τι αφορά το πώς οι πελάτες της ΕΤΕΠ μπορούν να ασθενιστούν ε, κάποιους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους. Είναι θέμα προθυμίας. Καταρχήν μπορούμε να έχουμε αυτούς τους όρους στις συμβάσεις που υπογράφει η ΕΤΕΠ ε, με τους πελάτες της. Ή αυτά τα κριτήρια να τα περάσουμε στους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς μέχρι να φτάσουν στους τελικούς δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΤΕΠ και όταν οι ΤΕΠ και άλλες δημόσιες τράπεζες έχουν πρόσβαση στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό, στο μέλλον με το InvestEU, στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσθέσει κάποιες διατάξεις στους κανονισμούς του, θέτοντας προϋποθέσεις και όρους για το πώς χρησιμοποιούνται τα δημόσια κονδύλια. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της βιοπικιλότητας και τη στάθμισμα του άνθρακα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να βρεθεί στον πυρήνα των μελλοντικών προοπτικών και του οδικού χάρτη για το κλίμα της τράπεζας. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να στηρίξουμε σχέδια και να μην βλάψουμε τη φύση και το περιβάλλον. Και αυτό μπορεί να το κάνει η τράπεζα για να συμβάλλει στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και στην προστασία της φύσης χωρίς να προσφύγει σε αυτά τα καινοτόμα εντός εισαγωγικών εργαλεία που είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας ό,τι αφορά την προστασία της φύσης. Και τέλος, για την ενέργεια, όντως έχουμε σφοδρές συζητήσει για τη οδότηση που κάνει η ΕΤΕΠ σε σχέδια για το φυσικό αέριο. Και πέρυσι ε, είχε μια πρωτοφανή πρωτοβουλία η ΕΤΕΠ, απαγορεύοντας τη χρηματοδότηση των ορεικτών καυσίμων και μέσω των χρηματοοικονομικών ε, διαμέσων. Βέβαια, Είπαμε ότι μέχρι το 2050 θέλουμε να έχουμε μια ουδέτερη οικονομία περιβαλλοντικά. Και αν συνεχίσουμε την δημόσια χρηματοδότηση των ορεικτών καυσίμων, ποτέ δεν πρόκειται να το καταφέρουμε. Επίση, έχουμε και οικονομικά επιχειρήματα. Ε, σήμερα οι τράπεζε ε, αν επενδύουν σε αγωγού φυσικού αερίου που έχουν 40-50 χρόνια ζωή ε, δεν συμφέρει, δεν είναι προσοδοφόρο οικονομικά. Οπότε είναι χαμένε επενδύσει θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα δημόσια κονδύλια να χρησιμοποιούνται για διορατικά σχέδια και όχι για την εφαρμογή συνταγών του παρελθόντος, που ήταν κάποια στιγμή χρήσιμες, αλλά όχι πια. Σας ευχαριστώ. Έχουμε σχεδόν εξαντλήσει το χρόνο μας, αλλά στο Catch δύο ε, συνάδελφοι μου ζήτησαν το λόγο και μια και προσφέρθηκαν να μείνουν λίγο παραπάνω οι διερμηνείς, θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό μόνο όμως στη διαδικασία του Catch the Eye στον Sven Giggold και μετά στον Mick Wallace. Ο Sven Giggold έχει το λόγο. Όχι, έχει χάσει τη σύνδεση του κύριο Giggold, οπότε μπορείτε να δώσετε το λόγο στον κύριο Wallace, τον επόμενο μιλητή. Ο Mick Wallace. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου απευθυνόταν στον συμπατριώτη μου, τον Ιρλανδό Άντριο Μακδάουελ. Είπα, ναι, είπαμε ότι θα χρησιμοποιηθεί για δάνεια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προκειμένου να φτάσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες. δημόσιες τράπεζες δεν έχουμε πια όμως στην Ιρλανδία. Πώς θα μερεμνήσουμε ώστε και οι ιδιωτικές τράπεζες να δίνουν χρήματα να δοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ιρλανδία, που είναι αυτές που τη χρειάζονται περισσότερο από οποιοδήποτε γιατί έχουν λιγότερα χρήματα, έχουν υψηλή ενεργεία, έχουμε και πρόβλημα τουρισμού και έχουμε και τους κανόνες ε, τήρησης αποστάσεων κοινωνικών. Όλα αυτά θα δυσκολέψουν τη ζωή πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. η κυβέρνηση βοήθησε στη διάρκεια της κρίσης ε, σημαντικά. Από τη στιγμή που θα ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις, οι προκλήσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες και η ζωή τους ακόμη πιο δύσκολη. Η ΕΤΕΠ, λοιπόν, όμιλος ΕΤΕ, μπορεί να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο και οι ενδιάμεση χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που χρησιμοποιεί να πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε τα χρήματα να φτάνουν πραγματικά σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ. Η ερώτηση αυτή απευθύνεται στους κυρίους Μακδόουελ και Μόλτερερ. Θα στείλουμε γραπτό στην ερώτηση στον κύριο Μακδόρελ, αλλά στον κύριο Μόλτερ μπορούμε να δώσουμε το λόγο για να απαντήσει. First of all... Πρώτα απ' όλα, ναι, επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο κύριος Σόλ. Ακριβώς, ό,τι αποφασίσαμε ισχύει για την κλιματική αλλαγή. Ο στόχος παραμένει 100% είμαστε προσιλωμένοι εκεί. Δεν νομίζουμε ότι η προσπάθειά μας για την πανδημία έρχεται σε σύγκρουση με τον στόχο που αφορά την κλιματική αλλαγή. Το θέμα του αξιόχρεου, το θέμα του Ταμείου Εγγύησης, όλα αυτά τα έχουμε επιστρατεύσει ανάλογα τι θα χρειαστεί και εννοείται ότι οι ΜΜΕ θα καλυφθούν από τις εγγυησει τα δύο τρίτα θα τους δώσουμε. Αλλά φυσικά και χρειάζεται να υπάρχει ενδιάμεσο όσον αφορά τη δανειοδότηση. Εθνικές τράπεζες, ε, τράπεζες, promotional εθνικές, ε, οτιδήποτε πλατφόρμα, οτιδήποτε χρειαστεί να συγκροτηθεί, ούτως ώστε να φτάσουν αυτά τα χρήματα στι ΜΜΕ. Μέχρι σήμερα ήταν πολύ θετική η εμπειρία μας με τους ε, ενδιάμεσους. Και όσον αφορά το φαντ και όσον αφορά την τράπεζα. Οι προποθέσεις είναι όπως έχουν ταχθεί από το Ταμείο. Θα διαβάσω φυσικά στον κύριο Αντιπρόεδρο όλα όσα ρωτήσατε. Η πρώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Οπότε, να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τους ομιλητές, τον κύριο Μόλκερ, τον κύριο Μικτάουρ, τον κύριο Παλέρμο και τον κύριο Σόλ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και από τις δύο επιτροπές, προϋπολογισμών και ε, ε οικονομικών τι ερωτήσει θα είμαστε σε επαφή και θα εξασφαλίσουμε ότι θα λάβει τι ερωτήσει σα, κ. Μακδάβολ, και θα σας ε, διαβιβάσει τι απαντήσεις. Και πάλι σας ε, ευχαριστούμε. Πέρας τη συνεδριάσεως. Δυσχερέστε.